Bien, chers collègues, nous allons euh, débuter. Je pense que certains collègues nous rejoindront. Euh, cet après-midi, notre session est... Λοιπόν, Θα μιλήσουμε για τη Λιβύη και πιο συγκεκριμένα στις εμπειρίες, στην εξέταση των εμπειριών, στα μαθήματα που έχουμε πάρει, εν πάση περιπτώσει, μετά από την στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, πέρυσι πλέον, χρονολογικά η προσπάθεια αυτή γίνεται ένα χρόνο, ακριβώς ένα χρόνο, μετά από τους πρώτους ευρωπαϊκούς βομβαρδισμούς στις 19 Μαρτίου. Διευκρινίζοντας βέβαια ότι από τις 19 Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαρτίου δεν ήταν τότε επιχείρηση του ΝΑΤΟ, ήταν μια ad hoc συμμαχική επιχείρηση και το ΝΑΤΟ ανέλαβε την ηγεσία της επιχείρησης μετά το τέλος του μηνός Μαρτίου θα de l'état-major Λοιπόν, προσπαθούμε καταρχάς βέβαια και αυτή είναι η δική μας δουλειά να μείνουμε στα πολιτικά συμπεράσματα και ιδιαίτερα τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η κυρία Γκόμες που είναι η συγγήτρια για τη Λιβύη και η οποία μαζί με τον κύριο Σαλαφράγκα επεσκέφθη τη Λιβύη ε, με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εδώ και ένα μήνα, για να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα εν πάση περιπτώσει για τους Ευρωπαίους, τι συνέπειες είχε η παρέμβαση για τη χώρα, τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφαλείας και θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα ακριβώς θα μιλήσουμε για τα βασικά λειτουργικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα της νατοικής επιχείρησης στη Λιβύη. Στρατηγέ μου, νομίζω ότι θα κάνετε μία προβολή ορισμένων διαφανειών. Εγώ για τη διάρκεια της προβολής θα, δεν θα κρύβω την οθόνη και μετά θα γίνει συζήτηση και θα τεθούν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω την παρέμβασή μου στην αγγλική γλώσσα και πριν επανέλθω στη γαλλική για να δώσω απαντήσεις, να διευκρινίσω λίγο το πλαίσιο της παρέμβασής μου, ένα πλαίσιο το οποίο εγγράφεται σε ακριβώς αυτή τη διαδικασία εκμετάλλευση των εμπειριών. Μια διαδικασία η οποία διεξάγεται, είναι εν εξελίξη. Τα συμπεράσματα λοιπόν τα οποία, στα οποία θα αναφερθώ είναι τα πρώτα που έχουν εντοπιστεί στα πλαίσια της επιχείρησης και είναι αντικείμενο προσεκτικής ανάλυσης ακριβώς για να γίνουν χρησιμοποιήσιμα σαν συμπεράσματα και να έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε τα μέτρα τα κατάλληλα για να καλύψουμε κάποιες αδυναμίες τις οποίες διαπιστώσαμε να βελτιώσουμε ό,τι χρήζει βελτίωσης. Ένα άλλο σημασιολογικό εκ των προτέρων σημείο που χρήζει διευκρίνηση είναι οι λεγόμενες capabilities, οι επιχειρησιακές ικανότητες. Αυτό για μας έχει μια ευρυτάτη έννοια. Δεν πρόκειται μόνο για εξοπλισμούς και για προγράμματα, αλλά και για, ε, ε, θέματα οργάνωσης, ε, για θέματα σκέψης, λογικής, και χρησιμοποιούμε τον αγγλικό όρο capabilities ή capabilities με ε, πολύ ευρύ ε, τρόπο. Λοιπόν τώρα θα ήθελα να σας ε, δώσω κάποιες διαφάνειες για αυτό που πιστεύουμε στο ΝΑΤΟ ότι ήταν τα βασικά μαθήματα αυτής της επιχείρησης. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τον προηγούμενο χρόνο την επιχείρηση Unified Protector. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικά πλαίσιο, νομίζω ότι πετύχαμε τους πολιτικούς στόχους και οδηγηθήκαμε σε μια επιτυχή γενικά επιχείρηση για τον ΝΑΤΟ. Πέραν όμως της επιτυχίας αυτής, η επιχείρηση Unified Protector, ενοποιημένος προστάτης, μας δίνει τη δυνατότητα για να δούμε ποια ήταν τα λάθη, ποια ήταν τα κενά, ποιες είναι οι ατέλειες που πρέπει να βελτιωθούν και να εντοπιστούν επίσης και οι βέλτιστες πρακτικές για χρήση στο μέλλον. Η παρουσίαση λοιπόν αυτή με αυτά θα ασχοληθεί, θα δούμε ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε από την επιχείρηση αυτή σαν ΝΑΤΟ για το μέλλον. Καταρχάς, το ΝΑΤΟ λειτουργήσε. Η επιχείρηση στη Λιβύη ήταν η πρώτη εφαρμογή της νέας στρατηγικής 2010. Η επιχείρηση αυτή έδειξε τη σημασία που έχει το ΝΑΤΟ στη νέα δυναμική ε, της ασφάλειας του περιβάλλοντός μας. Το ΝΑΤΟ στάθηκε ικανό να σχεδιάσει, να εγκρίνει και να εκτελέσει την αποστολή αυτή σε 14 ημέρες. Πέραν αυτού, οι κοινέ δομέ του, του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια του πολεμικού σεναρίου που περιλαμβάνει ναυτικέ επιχειρήσει και στα πλαίσια της πολυεθνικής συμμετοχής συμμάχων αλλά και εταίρων εκτός της συμμαχίας. Ήδη εξ αρχή βέβαια ασκήθηκε κριτική. Υπήρξαν διαφορές και αποκλίνοντα πολιτικά συμφέροντα ανάμεσα σε ορισμένες χώρες και αυτό φυσικά ήρθε στην επιφάνεια. Προσωπικότητες δήλωσαν ότι διαφωνούν με την επιχείρηση αυτή και τελικά μόνο λίγες χώρες πήραν μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως να πει κανείς ότι τη απουσία μιας μίζωνος απειλής για τη συμμαχία τα βασικά συμφέροντα των κρατών μελών δύσκολα καταλήγουν σε απόλυτα κοινούς κανόνες για το ΝΑΤΟ πέραν των επιχειρήσεων δεν υπήρξε ε, αναγκαστική αν θέλετε υποχρέωση όλων των χωρών να συνεισφέρουν. Και ορισμένες από τις χώρες του ΝΑΤΟ θεώρησαν ότι θα απέχουν. Τέτοιες αποφάσεις δεν επηρεάζουν βέβαια τη συνένεση, αλλά στερούν τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης για το ΝΑΤΟ δεν θα ήθελα αυτό να ερμηνευθεί ή να παρερμηνευθεί σαν αδυναμία της συμμαχίας. Η συμμαχία είναι ικανή να διαχειριστεί τη συνενετική βάση επί της οποίας βασίζεται η αντίδρασή του ανεξαρτήτως των διαφορετικών αντιλήψεων, συμφερόντων και παρουσιάσεων του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης. Ένα άλλο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η εμπλοκή των εταίρων ήταν κομβικό σημείο για την επιτυχία της επιχείρησης. Η επιχείρηση αυτή επικύρωσε, θα έλεγα, το, θα έλεγα τον ρόλο των εταίρων, των χώρων που συμμετέχουν με διαφάνεια και έδωσε τη δυνατότητα στις χώρες που το επιθυμούσαν, στις πρόθυμες χώρες να πάρουν μέρος. Υπήρξε αποτελεσματικότητα σε τομέα πολιτικής στήριξης, συνειδητοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος, και κατανομή ε, και κυκλοφορία πληροφοριών. Η συμμαχία λοιπόν θα συνεχίσει τις προσπά... η συμμαχία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, όχι μόνο οι πέντε χώρες που είναι σε αυτή εδώ τη διαφάνεια, αλλά και άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη πολιτική στήριξη στο ΝΑΤΟ, θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις χώρες. Επιπλέον διαδραστικά και με την πολιτική αεροπορία και με την αυσιπλοεία θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχύσουμε την εικόνα που έχουμε στα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα στα πλαίσια της αραβικής του συνιστώσης. Λοιπόν, τώρα, εμείς αποδείξαμε ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το πρόβλημα. Η συμμετοχή πολιτικών, μη στρατιωτικών θα έλεγα, οντοτήτων εξ αρχής είναι κάτι το ευεργετικό και σε επίπεδο προγραμματισμού και σε επίπεδο εκτέλεσης και τώρα μετεγχειρητικά σε εισαγωγικά συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία δράσης των Ηνωμένων Εθνών όπως επίσης και με τον Ερυθρό Σταυρό. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία κυρίως και στηρίζει ε, τις ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, αλλά από μόνο του δεν είναι σε θέση να δώσει μια πλήρη απάντηση σε σχέση με τους στόχους τους οποίους έχει θέσει και εξαρτάται από άλλους πολιτικούς οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά το ΝΑΤΟ ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο και σε αυτή την πολιτική διάσταση. Οι περισσότεροι από εμά θα συμφωνήσουν ότι τίποτα δεν είναι καλύτερο σε επίπεδο επικοινωνίας από ότι η επιτυχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εξαιρετικές και στρατικές στρατηγικές επικοινωνίες. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων και λόγω του ότι η Λιβύη ήταν μια κρίση η οποία εξελισσόταν με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες και με εναλλασσόμενες συνθήκες επιτόπου, διαπιστώσαμε κάποια κενά τα οποία προσπαθήσαμε εκ των υστέρων να καλύψουμε στο επίπεδο της επικοινωνίας. Αλλά ε, ε, εξαπλώσαμε θα έλεγα συγκεκριμένες ικανότητες οι οποίες με επιτυχία μπόρεσαν να είναι αποτελεσματικές. Συνεχίζουμε εμείς να εξετάζουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής Χρειάστηκε να λειτουργούμε με βάση την αρχή της πρόληψης, να αντιμετωπίζουμε θέματα πριν γίνουν απόλυτα γνωστά από τα μέσα ενημέρωσης, να καλύψουμε τα κενά αξιοπιστίας τα οποία μπορεί να είχαμε στην αρχή της επιχείρησης, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον τομέα της ενημέρωσης καταστήσαμε τα μηνύματα του ΝΑΤΟ αποτελεσματικότερα. Τα μηνύματα αυτά είχαν και μακροπρόθεσμη επίδραση. Και η συμμαχία δεν μπορεί να, να περιοριστεί στην επιχειρησιακή της επιτυχία στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα πρέπει να συνεχίζει την εμπλοκή της και την παρέμβασή της στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει όθηση για να προχωρήσουμε στην επόμενη ε, κρίση ε, όπως θα την παρουσιάσουν τα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να αναφερθώ στη συλλογή πληροφοριών, τον έλεγχο, την εποπτεία, την αναγνώριση και τους στόχους, την δυνατότητα ε, στόχευσης την οποία είχαμε. Η έλλειψη δυνάμεων σε επίπεδο ξηράς κατέστησε απαραίτητο για τον ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει μια συνειδητοποίηση του θεάτρου των επιχειρήσεων η οποία να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε στοιχεία αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών υπτάμενα. Ταυτόχρονα και μετά από τις πρώτους βομβαρδισμούς οι αντίπαλες δυνάμεις άλλαξαν τακτική και αναγκαστήκαμε και εμείς να προσαρμόσουμε την δική μας τακτική και να προσαρμοστούμε ε, σε μια κατάσταση ε, η οποία πολλές φορές ε, έβρισκε τους αντιπάλους μας να κρύβονται σε περιοχές με πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού. Το ISR λοιπόν, η ικανότητά μας αυτή όπως βλέπετε εδώ μπροστά μας δείχνει τι εύρος μέσων χρησιμοποιήσαμε ε, δείχνει επίσης και το προσωπικό το εξειδικευμένο που είναι απαραίτητο για την εκμετάλλευση και διάδοση των αποτελεσμάτων αυτών των μορφών ελέγχου. Το ISR λοιπόν, αναγνώριση, στοχοποίηση κτλ. δεν είναι απλά ένας πολλαπλασιαστής ε, ικανότητας. Είναι κάτι το οποίο ε, είναι απαραίτητο για τη σωστή διεξαγωγή της επιχείρησης και τον προγραμματισμό. Θα πρέπει να δούμε όμως και με κριτικό μάτι το τι κάναμε. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι, ο Καναδάς και οι υπόλοιποι εταίροι ε, διέθεσαν τον περισσότερο εξοπλισμό. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι η επιτυχία της επιχείρησης εξαρτήθηκε επίσης και από δυνατότητες τις οποίες μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείες μπορούσαν να μας προσφέρουν σε αυτή την κλίμακα. Είναι απαραίτητο λοιπόν για το ΝΑΤΟ να είναι βέβαιο ότι τέτοιου είδους δυνατότητες θα είναι περισσότερο διαθέσιμες και στην ίδια τη συμμαχία στο μέλλον. η ικανότητα να συγκεντρώσουμε μέσα ακριβώς συλλογής πληροφοριών στο μέλλον θα λειτουργήσει αρνητικά σε επίπεδο αποτελεσματικότητας της δράσης των δυνάμεων φιλικών ή όχι. Και θα μειώσει επίσης και τις δυνατότητες τις επιθετικές τις οποίες έχει το ΝΑΤΟ. Θα περιορίσει επίσης και την δυνατότητα να έχουμε μια κοινή συνολική αντίληψη του θεάτρου των επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο θετικός προσδιορισμός, οι προτεραιότητες, και το BDA, εκτίμηση δηλαδή των στόχων που έχουν, ε, ε, που έχουν χτύπηθει, είναι απαραίτητο ε, για την επανάληψή τους με μεγαλύτερη επιτυχία. Η έλλειψη επίσης εξειδικευμένου προσωπικού και η περιορισμένη ίσως αρχιτεκτονική ανταλλαγής πληροφοριών που λειτουργεί στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ έχει αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να συγκεντρώσει την προσοχή και τις επενδύσεις σε όλους τους ζωμείς όπου απαιτούνται ζωτικές επενδύσεις, όπως θα έλεγα αποθέματα βομβών τηλε, τηλε, ε, τηλεκατευθυνωμένων με ακρίβεια και τώρα βέβαια σε αυτή τη φάση της οικονομικής λιτότητας είναι δύσκολο οι χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις ικανότητές τους μεμονωμένα για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους απαιτήσει στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν το ΝΑΤΟ και η προσπάθεια και η ικανότητα που έχει το ΝΑΤΟ για τον έλεγχο εκ του αέρος των, ε, των ε, πεδίων των επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα της άμυνας με έξιμο τρόπο συνεργαζόμενοι η μία χώρα με την άλλη και με μεγαλύτερη ευελιξία. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τους στόχους μας, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί όπου μπορούμε να παράξουμε προστιθέμενη αξία, όχι μόνο σε επίπεδο όπλων αλλά και σε επίπεδο επιμελητίας. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στις ελάχιστες παράπλευρες απώλειες τις οποίες πετύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Οι πολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι ίσχυσαν εξ αρχής και η προσδοκία την οποία είχαμε για μηδενικές παράπλευρες απώλειες, απώλειες αμάχων εννοώ, επηρέασαν σαφώς την επιλογή των επίγειων στόχων πέραν την εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών που έχουμε και των, ε, ε, και των όπλων ε, ακρίβειας τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ακολουθήσαμε μία τακτική συγκεκριμένη σε όλη τη φάση της επιχείρησης. Και σε επίπεδο τακτικής και σε επίπεδο στρατηγικής είχαμε συγκεκριμένη εικόνα και υπήρχε πάντα για το χτύπημα συγκεκριμένων στόχων μία εκ των προτέρων θα έλεγα αδειοδότηση μετά από την εξέταση πάρα πολλών κριτηρίων. 11.000 χτυπήματα υπήρξαν από πλευράς της συμμαχίας, χιλιάδες όπλα εκτοξεύθηκαν, όλα τηλεχειριζόμενα με ακρίβεια σε ορισμένες περιοχές στοχεύσαμε τμήματα ορισμένων κτηρίων σαν παράδειγμα. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας. Η επιλογή του ελαχίστου, της ελαχίστης, ε, ελάχιστης ισχύω του όπλου επελέγει κάθε φορά έτσι ώστε οι ε, συνέπειες της έκρηξης να είναι περιορισμένες. Κάναμε ε, ό,τι τεχνικά ήταν εφικτό για να ελαχιστοποιήσουμε τις παράπλευρες απώλειες, αλλά σε μια περίπλοκη πολεμική επιχείρηση ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να εκμηδενιστεί. Και θα ήθελα να καταλήξω στα συμπεράσματα της Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας η οποία δημιουργήθηκε <clears throat> από το Συμβούλιο ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι το ΝΑΤΟ έκανε μια επακριβέστατη στρατηγική επιχείρηση για να αποφύγει ε, παράπλευρες απώλειες και αναγνώρισε το στόχο που είχαμε σαν ΝΑΤΟ και γι' αυτό πήραμε όλες, όλα τα μέτρα που χρειαζόταν γι' αυτό. Μίλησα για το τι μαθήματα ε, βγάλαμε εμείς, τι συμπεράσματα βγάλαμε για το μέλλον. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε κάποιες από τις δυνατότητες που παρουσιάζονται τώρα στο ΝΑΤΟ και στη διεθνή κοινότητα. Τέλειωσε η επιχείρηση, παρόλα αυτά το ΝΑΤΟ συνεχίζει την μεταεπιχειρησιακή φάση και η επεξεργασία των εμπειριών και των μαθημάτων που κάνουμε και σήμερα και επίσης η βοήθεια προς το ναό της Λιβύης και ε, τις κοινωνίες της περιοχής. Προσκαλέσαμε λοιπόν εμείς στη Λιβύη στον Μεσογειακό Διάλογο και συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα για δράσεις οι οποίες ε, θα βοηθήσουν στην απόσυρση και την έκρηξη των όπλων που έχουν παραμείνει εκεί. Συνεργαζόμαστε και με τα μέσα ενημέρωσης όπου αυτό είναι απαραίτητο και έχουμε μάλιστα αποχαρακτηρίσει απόρριτα έγγραφα έτσι ώστε να διευκολύνουμε τις έρευνες των διεθνών σωμάτων για τα διάφορα στοιχεία που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Συνεχίζεται επίσης ε, η περιφερειακή διαβούλευση για την ασφάλεια της περιοχής. Αυτό περιλαμβάνει συζητήσεις για το πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες ε, της νότιας ε, ε, περιοχής της Λεκάνης τη Μεσογείου και όχι μόνο της Λιβύης. Συνεχίζουμε και στηρίζουμε τις προσπάθειες της, Αφρο... Αφρικανικής Ένωσης και την ανάπτυξη των στρατιωτικών της ικανοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα των αερομε... της αερομεταφοράς. Όπως είπα λοιπόν, <clears throat> η επιχείρηση αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να βγάλουμε συμπεράσματα για να τα εφαρμόσουμε στο μέλλον. Πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε με ευελιξία, να διατηρήσουμε υψηλές στρατιωτικές ικανότητες, να έχουμε προσωπικό με ειδικά χαρακτηριστικά και ειδική κατάρτιση. Γι' αυτό λοιπόν τα συμπεράσματα αυτή της προσπάθειας ε, θα δοκιμαστούν στην πρακτική και στα πλαίσια της νέας δομής ε, ηγεσίας, της νέας ηγετικής δομής του ΝΑΤΟ και σε σχέση με την ε, by με την ανάπτυξη των στρατιωτικών δομών και των πολιτικών δομών του ΝΑΤΟ. Κλείνω λοιπόν την σύντομη παρουσίασή μου και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να δώσω απαντήσεις σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ακούστε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ε, χωρίς να θέλω να μπω σε πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες γιατί ίσως αυτό δεν μας είναι δυνατόν γιατί δεν είμαστε και ειδικοί όλων των ε, πραγμάτων εδώ τα οποία περιγράφηκαν. Όσον αφορά την ικανότητα συγκέντρωσης πληροφοριών, αγνώριση και παρακολούθηση το ISR, ε, αναφερθήκατε στην, ε, στην, ε, στη δυνατότητα αυτή η οποία είναι αμερικανικής προέλευσης και χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών θα ήταν δυνατόν να εξελιχθεί αυτό το σύστημα. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα πράγματα σχετικά. Ε, ποια, ποιες ελλείψεις υπάρχουν στο επίπεδο της Ευρώπης ή των χωρών μελών σε σχέση με όλες αυτές τις ε, διαδικασίες του ε, ορισμού των στόχων. Τώρα, όσον αφορά τις παράπλευρες απώλειες, σύμφωνα με την, έκφραση που, την τρέχουσα έκφραση που χρησιμοποιείτε, είπατε ότι κρατήθηκε σε ένα χαμηλό, ελάχιστο επίπεδο. Ε, όσον αφορά τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το ΝΑΤΟ, ε, ποια είναι τα εργαλεία λοιπόν που έχει το ΝΑΤΟ στη διάθεσή του για να προχωρήσει αυτή την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και εκ των υστέρων, ούτω ώστε να κρίνει με έναν ακριβέστερο τρόπο την ακρίβεια αυτής της αξιολόγησης, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και ένα κομμάτι της νομιμότητας αυτών των επιχειρήσεων ε, κατά την εξέλιξή τους και εκ των υστέρων βασίζεται εδώ. Ιδού λοιπόν και ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Κύριος Κέλερμα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την, ε, ε, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ε, βεβαίως, ε, όταν ορισμένες ε, χώρες του ΝΑΤΟ ανέλαβαν την ηγεσία, ολοκλήρωσαν αυτές τις επιχειρήσεις με επιτυχία. Ωστόσο, είπατε ότι η επιτυχία εξαρτάται από τις δυνατότητες αυτές. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή Με ανησυχεί η ενδεχόμενη έλλειψη των πόρων του ΝΑΤΟ για μελλοντικέ επιχειρήσεις. Γιατί αν φανταστείτε ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να καθυστερήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα, ίσως για έξι μήνες, τι, θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η εικόνα κατά συνέπεια. Άρα λοιπόν στο μέλλον όταν το ΝΑΤΟ έχει να αντιμετωπίσει το δεχόμενο μελλοντικών επιχειρήσεων και ίσως δύο ή τριών επιχειρήσεων ταυτόχρονα, τι θα είναι πρακτικά εφικτό ούτω ώστε να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις προκλήσεις. Και με αυτήν την ερώτηση σχετίζεται το θέμα τη συμβολή της φοράς ορισμένων χωρών μελών του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα της Δανίας, του Βελγίου, που συνέβαλαν ε, πολύ σημαντικά με τις αεροπορικές τους δυνάμεις, ενώ η σφορά άλλων χωρών ήταν πιο περιορισμένη. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση, θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ε, Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΝΑΤΟ παρόλο που έχω κάποιες επιφυλάξεις, θα ήθελα να το ευχαριστήσω για το έργο του στη Λιβύη. Ως συγγήτρια εδώ του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του πολέμου και πήγα εκεί αρκετές φορές και πρόσφατα με τον πρόεδρό μας για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στη Λιβύη. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική επιχείρηση και πραγματικά ε, σώσαμε ζωές με αυτή την επιχείρηση. Και αυτό ήταν καθοριστικό. Και είναι ακριβώ αυτό το είδου η επιχείρηση με τι ελάχιστε παράπλευρε απώλειε που εκπληρώνει του στόχου του Συμβουλίου Ασφαλείας όταν κάλεσε για ανάληψη ευθύνη προκειμένου να παράσουμε προστασία των πολιτών ε, που διώκονται από την ίδια τους την κυβέρνηση. Μόλις ήρθα από τη Ρωσία που ε, παρακολούθησα τα τοπικά τηλεπτικά προγράμματα και που παρακολούθησα όλη αυτή την ε, προπαγάνδα η οποία λέει ότι οι παράπλευρες απώλειες ήταν τεράστιες, ενώ συγγνωρίζουμε γνωρίζουμε ότι δεν ήταν και όλοι οι πολίτες με τους οποίους εγώ σε επαφή μου ήταν περιορισμένε οι παράπλευρες απώλειες. Και επίσης ισχυρίζονται ότι ήταν μια επιχείρηση η οποία δεν ήταν για να, προκειμένου να εκπληρωθεί το έργο της ανάληψης ευθύνη, αλλά για να αλλάξει η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο ευθύ εξ αρχής ότι το καθεστώς του Καντάφη ήταν προφανώς ο χειρότερος εχθρός του ίδιου του λαού. Όχι μόνο για ό,τι έκανε τις προηγούμενες δεκαετίες, ε, με ό, και όλοι να θεροτυφλούν ε, συμπεριλαμβανόμενων και των Ευρωπαίων ε, και α δούμε και τι επιθέσει στην Ευρώπη, για παράδειγμα τη δισκοθήκη στο, Βερολίνο ε, και τι άλλε τρομοκρατικέ επιθέσει. Αλλά βεβαίω όταν ξεκίνησε η εξέγερση, ο ίδιο ο Καντάφη υποσχέθηκε στο λαό της Λιβύη Ζάγκα Ζάγκα, το οποίο σημαίνει να σκοτώνει τους πάντες όπου τους συναντήσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη λύση χωρίς ε, να ανατραπεί το, ο Καντάφη. Και αυτό ήταν πολύ προφανέ για το λαό τη Λιβύη. Δεν ήταν όμω αυτός ο στόχος της επιχείρησης, αλλά βεβαίω ήταν αναπόφευκτο ότι θα συνέβαινε. Και νομίζω ότι πράγματι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό έγινε χάρη στον αγώνα των ίδιων των ε, Λιβύων, των Λίβιων, συγγνώμη, οι οποίοι πολέμησαν δεν ήταν μόνο, δεν ήταν η ξένη παρέμβαση, ήταν οι ίδιοι οι Λίβοι οι οποίοι πολέμησαν σε αυτόν τον πόλεμο. Και εγώ μπόρεσα να το διαπιστώσω όταν πήγα το Μάιο στη Βεγγάζη και είδα ότι πώς ε, ε, δίδονταν οι πληροφορίες από τους ίδιους τους ε, Λίβιους που θα έπρεπε, ποιους θα έπρεπε να βομβαρδίσουν και όλοι με τα κινητά έπαιρναν τις πληροφορίες αυτές από τους Λίβιους και τους ε, διαβίβαζαν στο ΝΑΤΟ. Και πραγματικά το λέω γιατί πιστεύω όταν μια εξαιρετική επιχείρηση, βεβαίω ε, θλίβομαι για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ήδη έκανε μια έκκληση στις 10 ε, Μαρτίου ε, να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει. Δεν υπήρξε συμφωνία για την εκκίνηση της επιχείρησης, γιατί ακριβώς υπήρξε ε, διαφωνία από τη Γερμανία, η οποία απήχε μάλιστα στην, ε, κατά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο είναι το κατά την άποψή μου. Έστω και αν θέλαμε να γίνει η επιχείρηση αυτή υπό την ΚΕΠΑ, τώρα καταλήγω ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνω, να το κάνουμε, γιατί ε, προποτίθενται διάφορες αρνητικές ε, δυνατότητες, ικανότητες, το οποίο δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ με τα όσα είπετε, αυτές δεν είναι ικανότητες που μπορούν να αποκτηθούν εν μια νυχτή, αλλά προϋποθέτουν πάρα πολλά πράγματα, κατάρτιση, εξοπλισμό κλπ. Και μια προετοιμασία. Ε, και υπάρχει, βεβαίω υφίσταται ε, και δεν είναι δυνατόν να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους, ε, από άλλους χάρες όπως είναι και οι Ηνωμένε Πολιτείες αλλά συνειδητοποιώ, αλλά εν ώψη ε, τα όσα ζήτησαν, των όσων ζήτησαν ήδη οι Λίβοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν κάποιες σημαντικές ε, συνέπειες όσον αφορά την πολιτική άμυνας και ασφάλειας, όχι μόνο για την Λιβύη, αλλά και για μας όσον αφορά τον έλεγχο, για παράδειγμα, των συνόρων. Γιατί εδώ είναι η δική μας ασφάλεια που διακυβεύεται. Λοιπόν, το κατά πόσο αυτές, ε, έχουμε λήψεις στο επίπεδο αυτό, ε, θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά. Υπάρχει αυτή, υπάρχουν αυτά τα ελλείμματα ή όχι. Ε, στα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για την παρουσία σύσης. Εγώ δεν είμαι ειδική στην κατάσταση για τη Λιβύα για τη Λιβύη, συγγνώμη. Αλλά το αντισταθμίζει η κυρία Γκόμε, νομίζω, για τους υπολείπου, τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπή. Θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή, είναι πιο ειδική ερώτηση. Αναφερθήκατε στην πρώτη, στην πρώτη διαφάνεια για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέροντας ένα είδος αποκλειστικής σχέσης μεταξύ της ίδιας της επιχείρησης και των ε, ΜΜΕ. Ε, σας κατάλαβα καλά και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να συγκριθεί δεν θυμάμαι πολύ καλά, λέει η ομιλήτρια. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στατηγέ, καλώ ήρθατε ε, για αυτή την, ε, και σε ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ε, διερωτώ με πόσο χρήσιμη ήταν η ανάπτυξη των δυνάμεων από αέρος. Ε, νομίζω ότι οι περισσότερες πτήσεις έγιναν από το αεροδρόμιο του Charles de Gaulle, ξεκίνησαν από εκεί. Το ΝΑΤΟ έχει αρκετές μη αμερικανικές ε, ε, δυνατότητες ε, για, την, για τα αεροπλάνα. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι κάποια από τα όσα μας είπατε και κάποια από τα όσα είπαν οι συνάδελφοι δεν τα καταλαβαίνω καλά και γι' αυτό η ερώτησή μου. Αυτή αυτές οι παράπλευρες απώλειες όπως τις αποκαλούμε. 30.000 θύματα ήταν επίσημα, 30.000 άνθρωποι έτσι. Από το Μεταβατικό Συμβούλιο 40.000 αναφέρθηκε ως ο αριθμός των θυμάτων. Τι είναι αυτό, παράπλευρες απώλειες, μικρές παράπλευρες απώλειες, 40.000 άνθρωποι θεωρούνται μικρή παράπλευρη απώλεια. Πώς είναι δυνατόν αυτό και σε σχέση με την εύστοχη χρήση του πυρός, πώς γίνεται να έχουμε 40.000 ανθρώπους θύματα, θύματα των 11.000 βομβών και ε, ε, βομβών που ερήφθησαν κατά τις επιθέσεις. Αυτή η αποστολή, ή πώς να το πω, όπως και να το αποκαλέσουμε, που επανειλημμένα ως μεγάλη επιτυχία με διατυμπανισμούς ε, εορτάστηκε και σαν έλεγε κανείς ε, σε σχέση με ε, τα όσα είχαμε ως στόχο απλά και μόνο την αλλαγή του καθεστώτος. Μίλησα με πολλούς από την Αφρικανική Ένωση και με εκπροσώπους και της κυβέρνησης και της Νότιας Αφρικής που και αυτοί πιστεύουν ότι αυτή η εντολή δεν έπρεπε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων να δοθεί και θεωρούν ότι αυτή η εντολή δεν μπορεί να ταιριάξει με το στενότερο πλαίσιο ή πνεύμα της εντολής για την προστασία των αμάχων. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να είναι συμβατό με τέτοιες επιθέσεις. 40.000 νεκροί άνθρωποι, 40.000 θύματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της προστασίας του πληθυσμού. Έτσι το κρίνετε εσείς. Και ποια συμπεράσματα μπορείτε να συνάξετε εσείς από αυτό την χρήση αυτών των επιθέσεων για το μέλλον. Αν όλα αυτά είναι τόσο επιτυχή όπως μας λέτε, τι συμβαίνει. Ζώνες απαγόρευσης πτήσεων ή ζώνες προστασίας των αμάχων στο μέλλον με το ίδιο, την ίδια διεύρυνση της εντολής θα έχουν πάλι τόσα θύματα στο μέλλον. Αυτό είναι το νόμιμο συμπέρασμα όσον αφορά την προστασία των ε, αμάχων. Η εντολή λέγεται protector. Η ίδια η εντολή Προστασία, προστασία του πληθυσμού. Αυτή είναι η προστασία που φαντάζεστε και που νομίζετε ότι είναι ιδανική. Και πάλι να θέσω το ερώτημα, κατά πόσον αυτό είναι μέρος της επιτυχίας με την κατάσταση που έχουμε σήμερα μπροστά μας ενώπιον των οφθαλμών μας στην Λιβύη. Διότι πολλά πράγματα από αυτά τα οποία ακούω είναι πολύ, ακούω, είναι πολύ ανησυχητικά. Σοβαρότατοι τραυματισμοί που από ένα άλλο καθεστώς ε, προκαλούνται από ό,τι από το προηγούμενο. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με αυτή την αποστολή. Στέφθηκε με επιτυχία αυτό, πιστεύετε. Κατά τα άλλα θα ήθελα έναν σαφέστερο ορισμό αυτής της έννοιας, σημασιολογικά, σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος και το κόστος το οποίο προκλήθηκε. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Στατηγέ, για την παρουσίασή σας. Καταρχήν θα ήθελα επίσης να πω ότι συμφωνώ με τα όσα είπε η Άννα Γκόμες, όταν μια ιδιαίτερα πετυχημένη επιχείρηση, αλλά ήταν μια αποτυχία παρόλα αυτά όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Νομίζω ότι εδώ χάσαμε τη μάχη στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το δικό μου ερώτημα αφορά τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των Ευρωπαίων Συμμάχων. Γιατί ακούσαμε και υπήρξαν πολλές φωνές που έλεγαν ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν συνέβαλαν με έναν σωστό τρόπο. Και γνωρίζουμε ότι ήταν καθοριστική η αμερικανική ε, εισφορά όσον αφορά την ανατροφοδότηση με καύσιμα των αεροσκαφών κλπ. και της ε, βάσεις απογείωσης των αεροπλάνων. Ε, η δεύτερη ερώτηση αφορά το τι είδους διδάγματα θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από την παρούσα κατάσταση στη Λιβύη, από την προσπάθεια σταθεροποίησης μετά από αυτή την παρέμβαση. Ποια είναι τα διδάγματα για τον προγραμματισμό στην εποχή μετά την σύγκρουση. Κατά την άποψή σας, Ποια είναι η δυνατότητα διεπιχειρησιακών ε, αποστολών ε, με τρίτες χώρες, όπως είναι το Κατάρ για παράδειγμα. Θα ήθελα να σχολιάσετε. Τέλος, άκουσα, ε, διάβασα μια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας όσον αφορά την ανάγκη διεξαγωγής ερευνών για τους ε, θανάτους αμάχων στη Λιβύη. Η Amnesty International λέει ότι πολλοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών και δεν υπήρξε απολύτως καμία αποζημίωση. Πώς θα μπορούσατε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ και τέλος ο κύριος Ζήμκε. Ναι, σας ευχαριστούμε για όλες τις ε, ε, πληροφορίες που μας δώσατε, γιατί είστε στρατηγικός και όχι πολιτικός. Θα ήθελα να συγκεντρωθώ σε κάποιες ερωτήσεις στρατιωτικής φύσεως. Θεωρώ ότι από στρατιωτική άποψη η επιχείρηση αυτή ήταν ιδιαίτερως πετυχημένη. Έγινε, προετοιμάστηκε τάχιστα και ολοκληρώθηκε επίσης γρήγορα αλλά θα ήθελα να θέσω κάποιες πιο συγκεκριμένες και λεπτομερικές ερωτήσεις. Πολύ γρήγορα οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ε, κατέκτησαν τον ενέργειο χώρο ε, και αυτή η επιτυχία φάνηκε πολύ γρήγορα. Ε, το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Γιατί τελικά η Λιβύη είναι μια χώρα η οποία είχε σχετικά σύγχρονα αεροσκάφη, είχε ένα σύγχρονο σύστημα αεροάμυνας. Αλλά τελικά ήταν, φάνηκε ότι ήταν αναποτελεσματικές οι αεροπορικές δυνάμεις των ε, Λίβιων. Άρα και το ΝΑΤΟ είχε κάποιες απώλειες. Άρα λοιπόν γιατί πιστεύετε ότι κατακτήσαμε πολύ γρήγορα αυτό τον εναέριο χώρο. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή. Είπατε στις ε, πληροφορίες που μας δώσατε ότι για τον εντοπισμό των στόχων τελικά αναπτύχθηκαν πάρα πολλά χερσαία όπλα από ξηρά. εκτοξεύτηκαν όπλα από ε, Και είναι αλήθεια ότι για να καταστραφούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να προσφύγει κανείς σε αεροσκάφη επανδρομένα ή μη επανδρομένα. Ε, ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η αναλογία, αν δούμε αυτές τις χιλιάδες επιθέσεων. Ποια είναι η αναλογία δηλαδή μεταξύ των ε, επανδρομένων αεροπλάνων ή αυτών που δεν είναι επανδρομένα. Γιατί αυτέ είναι κάποιε τάσει που διαφαίνονται αυτή τη στιγμή. Και η τρίτη και τελευταία μου ερώτηση είναι η εξή. Αυτή ήταν μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ, αλλά ευτυχώ το ΝΑΤΟ ε, επίση είχε τη συνδρομή άλλων χωρών. Και στο πεδίο αυτό έχουμε πάντοτε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη συνεργασία, ε, το συντονισμό ορισμένων ε, παραμέτρων, τεχνικής φύσεως για παράδειγμα. Ε, ξέρουμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα με τα σουηδικά αεροπλάνα στην αρχή. Και νομίζω ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα για, όσον αφορά την τροφοδοσία με καύσιμα αυτών των σουηδικών αεροπλάνων. στη βάση αυτών των επιχειρήσεων στη Λιβύη, Λιβύη μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Στρατηγέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, θα ξεκινήσω από τις δύο ερωτήσεις που μου θέσατε και ίσως αυτό θα με, επιτρέψει να απαντήσω σε κά, κάποιες άλλες ερωτήσεις που συνδέονται με αυτές για το θέμα. Αν, για να έλθουμε στο θέμα των δυνατοτήτων μας, ε, των, των δυνατοτήτων που, των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν ε, των Ευρωπαίων Συμμάχων. Καταρχήν υπάρχει εδώ το εξής θέμα. Τα ντρόν, ε, τα μη επανδρομένα αυτά αεροσκάφη, ε, κάποια, ε, αποτελούν ένα έλλειμμα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές δυνατότητες. Ε, και εδώ ήταν σημαντική η αμερικανική εισφορά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο όσον αφορά την ανισορροπία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Και θα έλεγα ότι αφού το ΝΑΤΟ έχει έναν στόλο το Airwalks για να εξασφαλίσει έγκαιρης ε, προειδοποίησης μπόρεσε να παράσχει μια επαρκή κάλυψη. Ε, αυτή είναι μια δυνατότητα λοιπόν του ΝΑΤΟ η οποία ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και την οποία χρησιμοποιούμε και στο Αφγανιστάν. Για τα ντρόν λοιπόν, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρα και θα έλεγα επίσης ότι αφορά την ικανότητα συγκέντρωσης πληροφοριών, αναγνώρισης και παρακολούθησης. Ε, πίσω από τα τρόν υπάρχει η επεξεργασία των πληροφοριών και υπάρχει η ανάγκη να υπάρξει ειδικευμένο προσωπικό για να γίνει επεξεργασία όλου αυτού του όγκου των πληροφοριών, οι οποίε συλλέγονται και τι οποίε θα πρέπει να μεταδέψουμε σε κάποιε συγκεκριμένε ε, πληροφορίε, σε θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ειδικευμένο καταρτισμένο προσωπικό όσον αφορά την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών. Πρέπει να μετατραπούν συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, εδώ συνέβαλαν σημαντικά οι Αμερικανοί όσον αφορά την, ε, το προσωπικό και τη συνεχή ε, τακτική επεξεργασία του, των πληροφοριών για να υπάρχει μια συνεχή τροφοδοσία με αυτό το υλικό. Ε, θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τις πληροφορίες αυτές ε, χρησιμοποιούνται όλοι οι εθνικοί διάβλοι. Τρίτον, τρίτο σημείο που θεωρώ ότι είναι ουσιώδες είναι το ζήτημα του targeting και très précise Σωστή στοχεύση. Και εδώ προποτίθεται μια σωστή κατάρτιση, άρα ένα επαρκές προσωπικό, ούτω ώστε να υπάρχει κάλυψη επί 24 ώρες κατά τη διάρκεια όλων των επιχειρήσεων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι Αμερικανοί όσον αφορά το προσωπικό της, σωστή της σωστής στόχευσης ε, είναι απολύτως ε, επαρκές και μπορούν να αντισταθμίσουν τα δικά μας λύματα, τα λύματα των Ευρωπαίων σε αυτό το επίπεδο. Είδω λοιπόν αυτά τα τρία σημαντικά στοιχεία στο επίπεδο αυτό. Όσον αφορά τι παράπλευρε απώλειε, ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα εδώ. Ε, όσον αφορά τη διαδικασία, μου πρόκειται για μια διαδικασία και είναι η αυστηρότητα τη εφαρμογή αυτή τη διαδικασία, δηλαδή επιλογές οι οποίες έχουν ε, γίνει στο επίπεδο του προγραμματισμού όσον αφορά τους περιορισμούς για τις ε, επιθέσεις, του βομβαρδισμούς σε σχέση με τη φύση των στόχων. Άρα λοιπόν ευθύ εξ αρχή από το πάνω μέρος ε, της αλυσίδας σε πολιτικό επίπεδο μέχρι τον πιλότο που κάθεται στο αεροσκάφος όλα αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με αυτή τη διαδικασία. Και η αυστηρότητα της διαδικασίας αυτής επιτρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι λεγόμενες παράπλευρες απώλειες. Άρα λοιπόν Πρόκειται για ένα θέμα ε, διαδικασίες που ακολουθείται και επαρκούς κατάρτιση των πιλότων. Γιατί αυτό προϋποθέτει πραγματικά μία νοημοσύνη, μία ευφία αντίδρασης σε και, και, ταχύτητα όσον αφορά την απόφαση του να χτυπήσει κανείς, να βοηθήσει κανείς ή όχι. Και αυτό μάλιστα έχει γίνει κατά επανάληψη. Ε, τώρα, όσον αφορά τεχνολογία, αυτό το ανέφερα ήδη. Ε, πρόκειται για λέιζερ ε, που για, μεθόδους, για συσκευές λέιζερ που καθοδηγούν τις ε, βόμβες και που παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια για να μείνει κανείς στην ακτίνα που, έχει κανείς, ε, που επιθυμεί κανείς εκ των προτέρων, ούτως ώστε οι συνέπειες της έκρηξης να μην υπερβαίνουν αυτό την ακτίνα. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερο σημαντικό και σε συνάρτηση με τη φύση του στόχου ε, γίνεται μια, σχετική, μια αντίστοιχη προσαρμογή χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτό το μοντέλο ε, Ιδού λοιπόν, ε, εξού και η σημασία να έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα όπλα, τις συγκεκριμένες βόμβες. Άρα λοιπόν η διαδικασία καθώς εκ των προτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αλλά και στη ε, μετέπειτα φάση γιατί χάρη των ηλεκτρονικών μέσων που βρίσκονται στο αεροσκάφος γιατί είναι τα αεροπλάνα αυτά ε, θα μας επιτρέψουν να, κάνουμε, να προβούμε στην αξιολόγηση μετά τον βομβαρδισμό με την ακρίβεια που απαιτείται γιατί όλα αυτά ε, κινηματογραφούνται. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η οπτικοποίηση και επιτρέπει αυτή την αξιολόγηση εκ των υστέρων. Δεν υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση μιας ε, βεβαίως ζημίας από, το να, από αυτή που γίνεται επί τόπου. Ε, ε, ε βεβαίως εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε το προσωπικό εκεί επί τόπου και χρειάστηκε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα αυτόν τον περιορισμό. Ε, και γι' αυτό, επειδή δεν είχαμε αυτό το προσωπικό εκεί, ε, προσπαθήσαμε να μειώσουμε ως το δυνατόν το περιθώριο των ασφαλμάτων. Να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο ακριβείς στους βομβαρδισμούς. Τώρα, όσον αφορά τα εργαλεία, υπάρχουν λοιπόν τα όπλα που μας βοηθούν, τα πυρομαχικά που μας ε, ε, βοηθούν. Υπάρχει ο εξοπλισμός ο οποίος ε, επιτρέπει μία αξιολόγηση μετά την, τον βομβαρδισμό και επίσης όπως σας είπα η αυστηρότητα της διαδικασίας και η τήρηση των κανόνων και η ποιότητα κατάρτισης εκπαίδευσης των πιλότων γιατί οι περισσότεροι πιλότοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να είναι οι πιλότοι πρώτης ε, γραμμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξεκινήσω με τις παράπλευρες απώλειες γιατί αυτό ε, συνδέεται με κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια. Βεβαίως θα παραμείνω εδώ στο στρατιωτικό πεδίο. Δεν θα επισέλθω σε πολιτικά ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να παναλάβω ότι οι παράπλευρες απώλειες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες στη Λιβύη και θα ήθελα να, να δείτε την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα αυτό ακόμα και την έκθεση της ε, Διεθνούς Αμνηστίας που μόλις είδε το φως. Ο αριθμός των θυμάτων υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένος και δεν μπορώ παρά να σας ζητήσω να προσέξετε σε αυτά τα δύο, τα δύο έγγραφα τα οποία ε, δεν είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικά του ΝΑΤΟ ούτως ή άλλως, αλλά αναγνωρίζουν παρόλα αυτά το τι έγινε, το έργο που έκανε. Τώρα για να επανέλθω στο θέμα των ε, δυνατοτήτων και των μελλοντικών του δυνατοτήτων. Κατά πόσο το ΝΑΤΟ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μελλοντικές επιχειρήσεις. Δεν, ε, βλέπω, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά ποια είναι ε, τα ποιοι είναι οι λόγοι που πίσω από την ερώτησή σας. Γιατί για μένα το επίπεδο των φιλοδοξιών του ΝΑΤΟ παραμένει το ίδιο έτσι όπως διατυπώθηκε στη Λισαβόνα. Και ένα δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να μας κάνει να εξετάσουμε το δεχόμενο μιας αλλαγής είναι οι δηλώσεις που έγιναν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με έναν στρατηγικό αναπροσανατολισμό των Ηνωμένων Πολιτειών ενδεχομένω, αλλά αυτός ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός ε, δεν ε, μπορεί να παρακάμψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, ε, αν θέλουμε να ε, ξαναγίνει μια επιχείρηση unified, του τύπου Unified Protector τους προσεχούς μήνες, ε, κατά την άποψή μου θα γινόταν με τον ίδιο τρόπο, θα υπήρχαν οι ίδιοι παράγοντες επιτυχίες και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες αδυναμίες. Εάν αυτό γινόταν την επόμενη χρονιά, ενδεχομένως τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί τον επόμενο χρόνο θα ξεκινήσει η μεταρρύθμιση των ε, δομών μας, η οποία αντλεί κάποια διδάγματα από τη Λιβύη, ιδιαίτερα στον φάτη σε και νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση όσον αφορά τον ε, έλεγχο και την... Ε, ε, και την δίκηση των επιχειρήσεων. Τώρα, θα έλεγα ότι έχει επιτευχθεί μια ε, ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Όπως σας είπα, η εισφορά των ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά την ικανότητα συγκέντρωση πληροφοριών, αγνώριση και παρακολούθηση στο ISR, αλλά από την άλλη οι Ευρωπαίοι ήταν ιδιαίτερως παρόντες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με τη στενή έννοια, όσον αφορά τις, ε, τους βομβαρδισμούς ιδιαίτερως, αλλά επίσης όσον αφορά την ε, δυναμική εξέλιξη των ίδιων των επιχειρήσεων, γιατί είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί οι οποίοι ε, υπήρξαν οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι πρόφησαν ε, τα πράγματα. Ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων είναι η... τα ελικόπτερα που ήταν δεδηλωμένη πρόθεση των ευρωπαϊκών χωρών να συμμετάσχουν τα ελικόπτερα τα οποία συνέβαλαν σημαντικά όσον αφορά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν στο επίπεδο της στόχευσης και της συγκέντρωσης επεξεργασίας των πληροφοριών εδώ ήταν σημαντική η αμερικανική εισφορά παρόλο που και οι Ευρωπαίοι εδώ συνέβαλαν, αλλά όσον αφορά την ανάπτυξη των δυνάμεων και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων υπό τη στενή έννοια, θεωρώ ότι εδώ ήταν καθοριστική η ευρωπαϊκή συνδρομή. Όσον αφορά τώρα τα αεροπλανοφόρα. Όσον σε σχέση με τον Unified Protector ε, είχαν το όνομα Σικελία. Very stable, very stable. Η Κρήτη. Και ε, υπήρχαν ε, πολλά αεροσκάφη και τα περισσότερα από τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ ε, ξεκίνησαν από την Σούδα, από την Ελλάδα ή από την Ιταλία και θα μπορούσα να σας πω επειδή αναφερθήκατε στο αεροδρόμιο του Charles το Charles de παρέμεινε υπό εθνική διοίκηση. Ποτέ δεν ε, πήχθη στην δίκηση του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή απογειώνονταν τα αεροπλάνα. Ε, περνούσαν μετά στην ε, δίκηση του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν οι βασικές βάσεις αυτές της Ελλάδας και της Ιταλίας. Euh, euh, λοιπόν, για το μέλλον, τι μαθήματα πήραμε, αν κατάλαβα, για το τι θα γίνει με τη Λιβύη στο μέλλον. Η κατάσταση ως έχει στη Λιβύη εξαρτάται και από τους ίδιους τους Λίβιους και από τη διεθνή κοινότητα. Είναι θέμα πολιτικό σε αυτή τη φάση, στο οποίο εγώ δεν θα επεκταθώ. Το θέμα των ε, δυνατοτήτων των στρατιωτικών που θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε σωστά τα σύνορα, αυτό νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με αυτά τα οποία είπα προηγουμένως με το ISR, με τη συλλογή πληροφοριών. Απαιτείται ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε τα χιλιάδες χιλιόμετρα που χωρίζουν τη Λιβύη από τους γείτονές της, σε περιοχές ιδιαίτερα ασταθείς. Εκεί πράγματι τα μέσα ενημέρωσης, ε, μέσα ελέγχου μάλλον εποπτείας είναι απαραίτητα και πρέπει πολλά να γίνουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις πιο ευαίσθητες περιοχές. Δεν νομίζω ότι το θέμα α, τίθεται με τον ίδιο τρόπο και στις υπόλοιπες χώρες. Για την λεγόμενη διαλειτουργικότητα με το Κατάρ και με άλλες χώρες. Δεν σημείωσα εγώ προβλήματα σε σχέση με τους Σουηδούς. Έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ίσως να υπήρξαν κάποια προβλήματα διαλειτουργικότητα στην προμήθεια καυσίμων. Πάντως είδα ότι δουλεύουν πολύ σοβαρά και ακριβώ η Επιτροπή Επιμελητίας προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στον τομέα των καυσίμων με τις χώρες του Περσικού κόλπου είτε τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε με το Κατάρ έχουμε το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιούν στρατιωτικό υλικό, συγγνώμη, είτε αμερικανικό είτε ευρωπαϊκό. Οι περισσότερες από τις χώρες αυτές έχουν επίσης μια εκπαίδευση στρατιωτικές τους δυνάμεις που περνούν από ε, στρατιωτικές σχολές είτε αμερικανικές είτε ευρωπαϊκές. Υπάρχει λοιπόν ένα επίπεδο διαλειτουργικότητας δεδομένο και ενδιαφέρον. Το δεύτερο σημείο και για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά τους και την δυνατότητα εκμετάλλευσης των μέσων τους, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο ε, καθοδηγήθηκαν από άλλες χώρες, το Κατάρ από τη Γαλλία, τα Εμμυράτα από τις Ηνωμένε Πολιτείες, εταίρους δηλαδή με τους οποίους έχουν πιο στενές σχέσεις από ότι με το σύνολο της συμμαχίας και γι' αυτό η ενσωμάτωσή τους έγινε με σωστό τρόπο. Υπάρχουν πολλά που μένει να γίνουν βέβαια ακόμα εδώ και γι' αυτό ακριβώς εμείς θέλουμε να πείσουμε τις χώρες αυτές να συμμετέχουν στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις χώρες αυτές σαν μελλοντικού εταίρους και για επιχειρήσεις στο μέλλον. Το θέμα των αντισταθμίσεων. Τι εννοώ εδώ. Είναι πολιτικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται αντικείμενο αντιμετώπισης από τις αρχές της Λιβύης και δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία να σας πω τι γίνεται στο Αφγανιστάν ίσως. Στο Αφγανιστάν και εκεί τίθεται το θέμα. Κάθε κράτος εφαρμόζει τους δικούς του δικούς της κανόνες στην περίπτωση αντισταθμίσεων ή αποζημιώσεων μετά από παράπλευρες απώλειες. Υπάρχει βέβαια σε επίπεδο γενικού στρατηγίου στο Αφγανιστάν μια σύσταση έτσι ώστε όλες οι χώρες να έχουν συστήματα αποζημίωσης των οικογενειών των θυμάτων. γιατί μια τόσο γρήγορη κατάκτηση του ενερίου ελέγχου. Γιατί η πολεμική αεροπορία του Καντάφη δεν ήταν και τόσο εκπαιδευμένη όσο πιστεύαμε. υπήρχαν προβλήματα συντήρησης ενός τμήματος του αεροπορικού στόλου. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά ίσως και γιατί η προηγούμενη επιχείρηση, Odyssey Down, έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά για την εξουδετέρωση των αντιεροπορικών δυνάμεων της Λιβύης. και γιατί τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ δούλεψαν καλά και λειτουργήσαν πράγματι αποτρεπτικά απέναντι στις δυνάμεις ε, του Καντάφη. Αυτοί οι τρεις παράγοντες εξηγούν τον απόλυτο έλεγχο της ζώνης με τέτοια ταχύτητα. Τα ποσοστά ανάμεσα σε μη επανδρομένα και σε επανδρομένα αεροσκάφη. Εδώ μιλάμε για 100% επανδρομένα και ε, τα μη επανδρομένα χρησιμοποιήθηκαν μόνο για φωτογραφίσεις, αναγνωρίσεις φωτογραφίσεις. Η διαλειτουργικότητα στο μέλλον, έχω απαντήσει νομίζω σε αυτό. Υπάρχει μια πραγματική βούληση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ να επιμείνουμε στο θέμα της διαλειτουργικότητας Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Connected Forces Initiative. Βασικό στόχος είναι η επίτευξη περισσότερης διαλειτουργικότητας όχι μόνο μέσα στους ε, συμμάχους αλλά και με ε, τους υπόλοιπους εταίρους. Η Λιβύη πράγματι ήταν ένα σημαντικό πεδίο θα έλεγα και συναντήσαμε ένα επίπεδο διαλειτουργικότητας το οποίο δεν αναμέναμε με ορισμένους εταίρους αλλά θα πρέπει να παραδεχθούμε επίσης ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να είμαστε πλήρως διαλειτουργικοί. Και θα τελειώσω για την ερώτηση για τα μέσα ενημέρωσης, αυτό το exclusive relation στο οποίο αναφέρθηκα. Δεν θα πρέπει να υπάρξει παρανόηση πάνω στον όρο τον οποίο χρησιμοποίησα. Ίσα ίσα θα πρέπει να κατανοηθεί με τον αντίθετο τρόπο, με την αντίθετη έννοια, ότι δηλαδή στην αρχή η δυσκολία του ΝΑΤΟ ήταν να ε, έχει προσωπικό στη διάθεσή του που να ασχολείται αποκλειστικά με τα μέσα ενημέρωσης. Στην αρχή ακριβώς, γιατί μετά οι διάφορες χώρες ε, κάλυψαν το κενό, αλλά στην αρχή είχαμε μια έλλειψη θα έλεγα ειδικών στο επίπεδο της επικοινωνίας όχι μόνο στις Βρυξέλλες, γιατί τα πράγματα δεν εξέλισσόντουσαν στις Βρυξέλλες, στην Άπολη, όπου υπήρχε το στρατηγείο και εκεί έπρεπε να γίνονται ανακοινοθέντα τύπου, να δίδονται και ένα τύπου κτλ. Θυμίζω ότι η πρώτη φάση ενημέρωσης έγινε στις Βρυξέλλες, αλλά μετά στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Και εκεί πράγματι χρειάστηκε να καλύψουμε κάποια κενά, γιατί υπάρχει ανάγκη ειδικών στην επικοινωνία που μας έθεσαν στη διάθεσή μας τα διάφορα κράτη-μέλη εκ των υστέρων μόνο. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Αν θέλετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνταγματάρχη μου. λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη στρατηγός λέει ο κύριος Ε, Πράγματι υπάρχει ένα ευαίσθητο όριο ανάμεσα, δυσδιάκριτο ανάμεσα στο πολιτικό και το στρατιωτικό. Euh, euh, λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση παιδαγωγικού πρακτικού τύπου για την ε, αλυσίδα διοίκηση, θα έλεγα κατά τη διάρκεια της ε, επιχείρησης από το πλοίο ή το αεροπλανοφόρο μέχρι το στρατηγείο, μέχρι το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Είπατε ότι όλα έπαιξαν ρόλο στα πλαίσια της ε, πρόσκτησης πρώτων και επικύρωσης εκ των των στόχων. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Μπορέσατε αυτήν την αλυσίδα ε, αλυσίδα είναι μερικές φορές πάρα πολύ μακρά. Βασίζομαι στην εμπειρία στρατιωτικών που μου λένε ότι από τις 19 Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαρτίου που ήμασταν σε μια ad hoc συμμαχία με συντονισμένα εθνικά στρατηγία επιτόπου, εκεί η ικανότητα δράσης μας ήταν ταχυτάτη ενώ όταν μπήκαμε στη διαδικασία ανάμεσα, εν πάση περιπτώσει, συνεργασίας του ΝΑΤΟ, Σμύρνη, Νάπολη κτλ, εκεί τα πράγματα δεν πήγαν τόσο γρήγορα. Ε, υπερβάλλω ή πράγματι υπήρξαν κάποια θέματα ως προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι ίσως δεν μπορείτε να μας δώσετε πάρα πολλές πληροφορίες ως προς αυτό. Η κυρία Κρόνμπεργκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη είναι πολύ ενδιαφέρουσα επειδή εκθέτει τις διαφορές σε σχέση με τις ικανότητες μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης. Μια από τις ερωτήσεις τώρα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινή Πολιτική Άμυνας είναι το pooling and sharing, η συνάθρηση και ο επιμερισμός ε, προσπαθειών και πόρων. Κάνουμε πολύ συχνά λόγο έχουν ε, και έχουμε χώρες και που έχουν ε, μειωμένες ε, δαπάνες άμυνας. Το pooling και sharing το βλέπετε ως μέρος της λύσης σε αυτό το πρόβλημα δυναμικού από πλευράς μας. Και η ερώτηση σε σχέση με τις δράσεις στη Λιβύη δίνουν κάποια μαθήματα ή κάποια παραδείγματα για αυτό το οποίο χρειάζεται για το pooling και sharing. Τι συμβαίνει σε σχέση με την εμπιστοσύνη, η έλλειψη εμπιστοσύνης για παράδειγμα όσον αφορά αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. I would like just to... Uh, Θα ήθελα, λέει η κυρία Γκόμες, απλά και μόνο να σχολιάσω αυτό το οποίο είπε η προλαλή για τις τους 30.000, 40.000 θύματα κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων. Πρέπει να σας πω δεν υποτιμώ καθόλου αυτό. Υπάρχει και πιθανότητα να είναι ακόμα υψηλότερος ο αριθμός των θυμάτων. Δεν θα έπρεπε όμως αυτά να αφορούν κατηγορίες κατά του ΝΑΤΟ. Διότι αυτό είναι το αποτέλεσμα του πολέμου που είχε ξεκινήσει ως εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των οπαδών του Γκαντάφη αν δείτε στην Σαχαουία, στην Μισράτα τι έγινε σε σχέση με την, το αδιάκοπο σφυροκόπημα όσον αφορά και την, ε, τις επιθέσεις των οπαδών του Γκαδάφη και τον εμφύλιο πόλεμο. Και αν δείτε <clears throat> και τους ε, όχι πολύ καλά καταρτισμένους Λίβιους στρατιώτες που πήραν τα όπλα με ό,τι είχαν στα χέρια τους για να καταπολεμήσουν αυτό το τυραννικό δολοφονικό καθεστώς. Δεν υποτιμώ καθόλου τον αριθμό των θύματων. Τα θύματα μπορεί να είναι ακόμα περισσότερα ίσως τελικά. Και όπως πρόσφατα αναφέρθηκε από τον ίδιο τον στρατηγό βλέποντας την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών και την πρόσφατη ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας που αναφέρει 53 ως θύματα της ε, δράσης ε, του ΝΑΤΟ. Είναι εκπληκτικό αυτό και γι' αυτό είναι τόσο ευγνώμονες ε, οι Λίβοι για αυτή, τη δράση. Αυτό είδαμε και αυτό η ίδια, η ίδια εγώ είδα και άκουσα και δεν θα σας έλεγα τίποτα παρά μόνο την αλήθεια όπως μου την ανέφεραν και οι Λίβοι σε σχέση με όσα είπε ο στρατηγός. Σαν αποτέλεσμα του πολέμου λοιπόν είχαμε και εξοπλισμό από τις δυνάμεις του Καντάφη που ήταν διάχυτος αυτός ο εξοπλισμός στην ε, περιοχή χημικά όπλα και ε, αντίστοιχος εξοπλισμός ε, πήγαμε στη Λιβύη σε αποστολή και είδαμε πρόσφατα ότι πολύ καλή δουλειά έχει γίνει ήδη για να εντοπιστούν και να βρεθούν αυτά τα χημικά όπλα και να αντιμετωπιστούν και ο εντοπισμός ε, αυτών των ε, ε, κρυψώνων και όπλων είναι σημαντική υπόθεση. Συμμετείχε το ΝΑΤΟ σε αυτή την προσπάθεια ή κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν να βοηθήσουν τους Λίβιους σε αυτή την προσπάθεια, μια και αυτοί δεν έχουν το πραγματικό δυναμικό για να το κάνουν μόνοι τους. Ευχαριστώ. Κύριο Στένοκ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Γκόμες έκανε λόγο για τα θύματα τον αριθμό 30-40 χιλιάδων που αφορά τον αριθμό των θυμάτων και είπε ότι οι ίδιοι οι στρατιώτες του Γκαντάφη, Λίβοι είναι αυτοί που προκάλεσαν τόσα θύματα. Πώς ήταν στρατιώτες και πώς ήταν μισθοφόροι, γιατί ακούμε τις πιο διαφορετικές φήμες ε, για τους μισθοφόρους. Ξεκινάνε από κάποιες εκατοντάδες και φτάνουμε σε μυριάδες. Ε και σε σχέση και με την ε, συμμετοχή αυτών των ε, μισθοφόρων που μάλλον αυτοί έκαναν τα πάνδυνα αντί για ε, τους ίδιους τους Λίβιους και για την προστασία του ίδιου του Γαντάφη μέχρι τέλους. Τώρα που έχει καταλαγιάσει ο ρημαδός να μάθουμε, να ακούσουμε τι έγινε με αυτούς τους μισθοφόρους. Συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν, ε, μπόρεσαν να επιστρέψουν στις χώρες τους. Τι συνέβη με αυτούς. Με ενδιαφέρει το θέμα των μισθοφόρων. Είναι όμως κάτι το εκπληκτικό όταν δεν είχαμε και ούτε ένα θύμα από πλευρά των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που να ε, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ε, εχθροπραξιών. Και θα ήθελα αυτό να μου το επιβεβαιώσετε αν πράγματι αληθεύει. Και μετά για την πληθώρα όπλων των, που κυρίως χρηματοδοτήθηκε από τους ίδιους από το Κατάρ το ίδιο. Ακούμε πολλά για αυτά τα όπλα, υπερβολικά πολλά όπλα που βρίσκονται και στα χέρια Ισλαμιστών ακραίων ε, αδυνάμεων που εξοπλίστηκαν αδιάκριτα και που ε, στη συνέχεια μπορούν να περάσουν στην ε, υποσαχάρια Αφρική, στη Δυτική Αφρική, στο Μαγκρέμπ και να δράσουν ως ακραίοι Ισλαμιστές. Έχετε κάποιες πληροφορίες και σε σχέση και με έναν από τους γιους, ε, γιους του Γκαντάφη ε, που ε, πήγε στην, στο, ε, στον Νίγηρα και σε σχέση με την δυνατότητα της, ας το πω έτσι, αποκατάστασης του προηγούμενου καθεστώτος. Κατά πόσον παίρνουμε σοβαρά τέτοιου είδους φήμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στρατηγέ. Έχετε εκ νέου το λόγο. με την αλυσίδα διοίκησης του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο στρατιωτικό εξοπλισμό μηχανισμό από τη μία και όλον τον πολιτικο-στρατιωτικό μηχανισμό από την άλλη που έχει έδρα στις Βρυξέλλες εδώ λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις στο εσωτερικό του Συμβουλίου, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, με φυσικά συμβουλές από πλευράς της Στρατιωτικής Επιτροπής της Συμμαχίας, που είναι θα έλεγα αυτός που ε, επιλέγει, ε, θα έλεγα, τις διάταγες και τα αιτήματα τα οποία το στρατιωτικό αρχηγείο της ΜΟΣ μεταφέρει στην Πολιτική Επιτροπή πριν δώσει μια διαταγή το στρατηγικό στρατιωτικό επίπεδο, θα πρέπει να περάσει από την Στρατιωτική Επιτροπή η διαταγή αυτή, η οποία θα γνωμοδοτήσει σε στρατιωτικό πάντα επίπεδο υπέρ του πολιτικού ε, οργανισμού, του Συμβουλίου δηλαδή, του ε, Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Και μόνο όταν συμφωνήσει το Συμβούλιο, τότε η διαταγή μπορεί να εκτελεστεί στα διάφορα ε, επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά. Μιλάμε το ΣΑΚΕΡ, το ανώτατο στρατηγείο, το ανώτερο στρατηγείο, το στρατηγικό επίπεδο δηλαδή, και μετά έχουμε το λεγόμενο λειτουργικό επίπεδο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν στην Άπολη, το οποίο απετελεί το από το ανώτατο στρατηγείο της Νάπολη, όπου υπάρχει και ο διοικητής της επιχείρησης, ο Force Commander, ο στρατηγός Μπουσάρ. Ο στρατηγός Μπουσάρ ήταν, θα έλεγα, αποσπασμένος στην διοίκηση του ΝΑΤΟ. Το στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις τρέχουσες επιχειρήσεις, ταυτόχρονα και για το κοσυφοπέδιο και πρέπει να διαχειριστεί και την καθημερινότητα χρειάστηκε να φύγει ένα κομμάτι του και να δημιουργηθεί ένα καινούριο πουλ της συγκεκριμένης επιχείρησης με βάση το προσωπικό της Νάπολης και με βάση ενισχύσεις αποσπασμένων από άλλα κράτη-μέλη ή από άλλες διοικητικές δομές του συμφώνου. Στη συνέχεια μπορείτε να καταβείτε ακόμα ένα επίπεδο μετά από το λεγόμενο λειτουργικό επίπεδο και φτάνετε σε αυτό που ονομάζουμε ε, τα διοικητικά κέντρα των συνιστοσών, μιας και δεν είχαμε ε, επίγειες δυνάμεις. Είχαμε λοιπόν ένα στρατηγείο αεροπορικών στρατιωτικών δυνάμεων, ένα ναυτικό, το οποίο βρισκόταν και αυτό στην Άπολη. Αυτή ήταν η αλυσίδα της διοίκησης, έτσι όπως υπάρχει σε μόνιμη βάση. Και αυτή είναι η δύναμη του ΝΑΤΟ ότι εκ των προτέρων δηλαδή είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε γιατί υπάρχει η αλυσίδα της διοίκησης και το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο μέσα από ασκήσεις έτσι ώστε να αναλαμβάνει τέτοιου είδους επιχειρήσεις αν και εδώ βέβαια πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις και είμαι βέβαιος ότι η μεταρρύθμιση της διοικητικής δομής θα βελτιώσει ακόμα την επιχειρησιακή ικανότητα της συμμαχίας. Τώρα αν είναι ε, θα έλεγα δίσκαμπτη ή βαριά αυτή η αλυσίδα της διοίκησης. Όταν είναι κανείς σε μια οργάνωση με 28 χώρες που παίρνουν αποφάσεις με συνένεση, δεν έχει κανείς την, δια, την αντιδραστικότητα, την άμεση εν πάση περιπτώσει αντίδραση που έχει σε άλλες περιπτώσεις όπως την επιχείρηση Odyssey Down. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχε συντονισμός ανάμεσα σε ορισμένες χώρες, υπήρχε μια εθνική δομή η οποία είχε προτεραιότητα στη λήψη των αποφάσεων, υπήρχε λοιπόν μια συγκεκριμένη θα έλεγα άμεση ανάγκη, αποδεδειγμένη και μια ανάγκη άμεσης αντίδρασης και εκεί έδωσαν τη λύση οι εθνικές δομές. Το ΝΑΤΟ δεν γίνεται αυτό, είναι προφανές ότι το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί έτσι. Και όπως είπα, θα πρέπει η απόφαση να λαμβάνεται σε επίπεδο 28 χωρών, θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει ξεκάθαρα, η διαδικασία να περνάει από όλη την αλυσίδα με τον σωστό τρόπο και οι διαταγές να έρχονται με την έγκριση του πολιτικού επίπεδου των 28 κρατών. Και αυτό απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο, ιδιαίτερα για να ξεκινήσει γιατί όταν ξεκινά μια επιχείρηση, εκεί θα έλεγα έχει κανείς την ίδια αντίδραση που μπορεί να έχει σχεδόν την ίδια σε μια εθνική στρατιωτική δομή. Σχεδόν, γιατί λέω σχεδόν. Υπάρχουν τα λεγόμενα εθνικά caveat, δηλαδή κάποια ειδικά εθνικά συμφέροντα. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα, τα τα συγκεκριμένα που έχει ο ένας και ο άλλος, η κάθε χώρα. Αυτό λοιπόν απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο. Όταν πρέπει να δώσουμε μια αποστολή σε ένα αεροσκάφος πρέπει να δούμε ποια χώρα είναι το αεροσκάφος γιατί μπορεί κάτι να κάνει και κάτι να μην μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Δεν μιλάμε για δύο-τρεις χώρες οι οποίες δεν έχουν κανένα θα έλεγα εθνικό κόλλημα να πάνε πιο γρήγορα. Αυτό που μπορώ να πω λοιπόν εδώ για να δείξω ακριβώς αυτή την αδυναμία, μια αδυναμία η οποία είναι και συνέπεια της δύναμης όμως. Η δύναμη του ΝΑΤΟ είναι η συνένεση των 28 χωρών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περνάμε από εκεί. Και το σύστημα επίσης των παράπλευρων απολειών είναι και αυτό αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της δομής. Λοιπόν, συνδυασμός και κατανομή. Είναι χρήσιμο. Γιατί όχι. Ιδιαίτερα στο σημερινό πλαίσιο. Τίθεται το θέμα της εμπιστοσύνης. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για την επιχείρηση αυτή στη Λιβύη. Σας μίλησα για τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης. Κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ εξοπλίζουν θα έλεγα τα αεροσκάφη αυτά με το προσωπικό τους, επανδρώνουν, συγγνώμη. Μία από τις χώρες δεν ήθελαν να υπάρχει προσωπικό της συγκεκριμένης χώρας. Οπότε έπρεπε επίσης να βρούμε προσωπικό για να συμπληρώσει τα κενά και το βρήκαμε. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να καλύψουμε τα κενά. Κατά τα άλλα δεν έχω κάποιο άλλο παράδειγμα να σας δώσω. Αναφέρθηκα στις καινοτομίες. Ένα νέο μέσο συλλογής πληροφοριών, το οποίο χρηματοδοτείται από 13 χώρες του ΝΑΤΟ, και το οποίο θα είναι μια συμπληρωματική ικανότητα α, της συμμαχίας. Θα είναι κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε στα πλαίσια της χρήσης αυτών των μέσων εάν πράγματι έχουμε εγγυημένη σαν ΝΑΤΟ πρόσβαση σε, αυτή, σε αυτό το μέσο, σε αυτή την ικανότητα. Αλλά καταρχάς έχετε απόλυτο δίκιο αυτό το οποίο μετράει είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε φίλους. Σχετικά λοιπόν, σχετικά λοιπόν με το Unified Protector, το συμβόλαιο αυτό θα έλεγα εμπιστοσύνη, εκτελέστηκε πλήρως. Οι Αμερικανοί όποτε χρειάστηκε να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους το έκαναν. Ενώ από την αρχή πήγαν στη δεύτερη γραμμή αν θα σε σχέση με την εξέλιξη της επιχείρησης. Ήταν παρόντες όμως αλλά ήταν εκεί. Λοιπόν, δούλεψε το πράγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για το pooling and sharing ξανά λοιπόν, εδώ ο Γενικός ε, Γραμματέας του ΝΑΤΟ επιλέγει πολιτικά αυτό το οποίο ονομάζουμε Smart Defense, έξυπνη άμυνα. Στόχος είναι όμως ένας, να επωφεληθεί κανείς από τις πολυεθνικές ε, ικανότητες για να αντισταθμιστούν οι εθνικές δημοσιονομικές δυσκολίες και να διασφαλίσει κανείς τις, οικονομι... τις ε, ικανότητες της στρατιωτικής δύναμης παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Αυτός είναι ο στόχος του Smart Defense. Σωστή ιεράρχηση των αναγκών, σωστή χρήση των εξειδικευμένων δυνάμεων. Σαν παράδειγμα η αστυνόμευση του εναερίου χώρου των βαλτικών χωρών. Κάποιες χώρες που έχουν την αεροπορική δυνατότητα καλύπτουν την ανάγκη αυτή υπέρ των χωρών των βαλτικών που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και οι βαλτικές χώρες εκεί βλέπουν ότι μπορούν να εμπιστευτούν τους συμμάχους της, γιατί εδώ και δέκα σχεδόν χρόνια οι σύμμαχοι συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή χωρίς ποτέ να αποστούν. Πάντως το κλειδί αυτού του συστήματος του πολυεθνικού το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε για να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας, κλειδί είναι η εμπιστοσύνη και η εγγυημένη πρόσβαση στις ικανότητες αυτές. Τώρα για τα συμπεράσματα τα στρατιωτικά μετά την αποστολή της Λιβύης και τι έχει απομείνει εκεί. Χημικά όπλα και συστήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν εκεί ή στον τομέα της εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας. Όχι, το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει σε αυτά. Οι χώρες του ΝΑΤΟ όμως μεμονωμένα σαφώς και εμπλέκονται μπορέσανε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα, όλες τις πληροφορίες που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Για τους μισθοφόρους δεν μπορώ να σας πω τίποτα εδώ. Πράγματι είναι γεγονός ότι υπήρχαν μισθοφόροι, τους οποίους πλήρανε ο Καντάφη, πόσοι ήταν δεν μπορώ να ξέρω. Θυμίζω ότι από πλευράς του ΝΑΤΟ δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός, ούτε καν τραυματίας λόγω πολεμικής ενέργειας. Τα όπλα τα οποία διέθεσε το Κατάρ ε, στους αντάρτες ήταν μια πρωτοβουλία του Κατάρ. η διαταγή δεν δόθηκε από το ΝΑΤΟ, δεν συζήτησε το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, η συνέλευσή του κάτι τέτοιο για τον εξοπλισμό των ε, Λιβύων ανταρτών. Το τι έγιναν τα όπλα αυτά ε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Είναι αλήθεια όμως ότι εξόπλισαν τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που πολέμησαν τις δυνάμεις του Καντάφη και βρίσκονται πάντα από ό,τι νομίζω τα όπλα στα ίδια χέρια η εκτίμηση την οποία κάνω για πιθανές απειλές από πλευράς του Ιού Καντάφη που έχει ε, καταφύγει στον Ήγυρα, νομίζω ότι εδώ κάνω μια προσωπική αξιολόγηση και δεν υπάρχει κανένας μα κανένας φόβος. Δεν υπάρχει καμία προοπτική. Ε, η εποχή Καντάφη ανήκει στο παρελθόν. Θα υπάρξουν νέες δυνάμεις αντιτιθέμενες ίσως, αλλά δεν θα υπάρξει μια εκ νέου επιστροφή της ε, φατρίας του Καντάφη. Μάλιστα, στρατηγέ μου, σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναλάβατε αυτό το μη εύκολο έργο. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία της εμπειρίας, εξολόγησης της εμπειρίας δεν έχει ολοκληρωθεί ε, και το σύνολο αυτής της διαδικασίας βεβαίως υπόκειται σε κάποιες ε, διπλωματικές ή πολιτικές ε, ερμηνείες στις οποίες δεν θελήσατε να επισέλθετε και ήταν αρκετά συνετό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που μας είπατε από στρατιωτική και τεχνική άποψη κάποια πράγματα και όλες αυτές τις αξιολογήσεις που θα είναι χρήσιμες για τις, Ευρωπα... για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστω και αν οι χώρες, και αυτό το επενθυμίσατε, έχουν ε, πάρα πολλές ε, κριτικές, ε, πάρα πολλές, πάρα ικανότητες και σκέφτομαι το, έργο, το δύσκολο έργο που εκτελούν οι πιλότοι των αεροσκαφών και επίσης θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι η συμμαχία δεν είχε κανένα νεκρό κάτι που πραγματικά είναι ανήκουστο για μια επιχείρηση τέτοια εμβέλεια. Και επίσης ε, νομίζω ότι μπορέσαμε μαζί με την Άννα Γκόμης να ε, διαπιστώσουμε το, την εμβέλεια και την ακρίβεια αυτών των βομβαρδισμών που πραγματικά ήταν υποδειγματική και, αν συγκρίνουμε με το Κόσοβο, η πρόοδος σε σχέση με την σωστή στόχευση ήταν πραγματικά σημαντική. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για αυτή την παρουσίαση και αυτή τη στιγμή οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Θα θέλαμε να μάθουμε τα συμπεράσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ στρατηγέ μου και θα ήθελα να σε υπενθυμίσω ότι σε 20 λεπτά στην Ολομέλεια για τα μέλη της Υποεπιτροπής και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ακούσουμε την κυρία Άστον, την ε, είπα, εκπρόσωπο, Επίτροπο Εξωτερικών Υποθέσεων.